Ε, Δεύτερη πληροφορία που έχω να σας δώσω. Ανησυχητικά νέα λαμβάνουμε από γειτονικές χώρες Μπαχρέιν, Συρία και Ιεμένη. Σε όλες αυτές τις χώρες οι διαδηλώσεις κατεστάλησαν και ήταν άνθρωποι αυτοί που διαδήλωναν για περισσότερη δημοκρατία και στρέφουν οι κυβερνήσεις τα όπλα κατά του λαού τους και οι κυβερνήσεις αυτές χάνουν κάθε ε, δημοκρατική νομιμότητα θα πρέπει να σταματήσει η βία και αυτοί που είναι υπεύθυνοι θα πρέπει ε, να ε, δικαστούν. Επόμενο θέμα προ ενημέρωσή σα. Αυτή την εβδομάδα η διεθνή κοινότητα γιορτάζει την εβδομάδα αλληλεγγύη με τις χώρες που πολεμούν τον ρατσισμό και την διάκριση με ε, βάση ε, τη φυλετική καταγωγή. Τελευταία πολλά έχουν γίνει στον ελεύθερο κόσμο για να εκριζωθεί ο ρατσισμός από την καθημερινή ζωή. Ξέρουμε ότι πολλά από μένου πρέπει να γίνουν και στα κράτη-μέλη και εκτός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Άλλο ένα θέμα προς ενημέρωσή σας. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα μάθαμε ότι ένας από τους συναδέλφους μας, ο κύριος Τάλερ, παρετήθηκε από τη θέση του στο Κοινοβούλιο και δεύτερος συνάδελφος, ο κύριος Στράσερ, και εκείνος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί από τη θέση του τις επόμενες μέρες. Τρίτο μέλος, ο κύριος Σεβερίν, αποχωρεί από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Και θα ανήκει στα μία εγγεγραμμένα μέλη πλέον. Αυτές οι παρετήσει είναι αποτέλεσμα σοβαρών καταγγελιών και κατηγοριών που εμφανίστηκαν στα μέσα ενημέρωσης για μη ε, σωστή, μη ορθή συμπεριφορά των μελών του Κοινοβουλίου. Σήμερα συνεκάλεσε εκτάκτο το Προεδρείο του Κοινοβουλίου για να συζητηθεί όλη η κατάσταση. Επίσης θα συνεδριάσουμε και σήμερα το απόγευμα για να συνεχιστεί η συνεδρίαση. Μιλώντα εκ μέρου ε, του Προεδρείου του Κοινοβουλίου και εκ μέρου της πλειοψηφίας των συναδέλφων του Κοινοβουλίου πρέπει να πω ότι είμαστε αποφασισμένοι να εφαρμόσουμε μια πολιτική μηδενικής ανοχής. Μηδέν ανοχή σε αυτού του είδους τις πράξεις που οδήγησαν στην παρέτηση των συναδέλφων μας. Σαν πρόεδρος εκλεγής από εσάς συνάδελφοι είμαι αποφασισμένος να διαφυλάξω την ειλικρίνεια και την τιμιότητα του Κοινοβουλίου και των μελών του Κοινοβουλίου. Έχουμε βαρύ βάρος, έχουμε μεγάλο βάρος στους ώμους μας ευθύνη γιατί μας εξέλεξαν οι πολίτες και μας έδωσαν την εξουσία να κυβερνήσουμε εν ονόματί τους και δεν θα πρέπει να προδώσουμε την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν. Το Προεδρείο αποφάσισε να μάθουμε το μάθημά μας από αυτά τα ατυχή συμβάντα. Το Κοινοβούλιο επιθυμεί ε, να πέσει άπλετο φως στα γεγονότα. Θα συνεργαστούμε με όλες τις αρμόδιες αρχές, ούτω ώστε να ρίξουμε φως σε όλα όσα συνέβησαν και να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε τις πληροφορίες που υπάρχουν. Το Προεδρείο μου ζήτησε να έρθω σε επαφή με Εθνικά Υπουργεία Εξωτερικών, τα Εθνικά Υπουργεία Εξωτερικών των μελών που προανέφερα, για να δούμε τι δράση ενδεχομένω θα αναλάβουν τα δικαστήρια των χωρών αυτών. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενισχύσει το δεοντολογικό του κώδικα όσον αφορά αυτές τις συμπεριφορές και θα πρέπει να είναι ε, πιο αυστηρές οι κυρώσεις που προβλέπονται για τέτοιες πράξεις. Οι πρόσφατες αυτές πράξεις, δράσεις έδειξαν την ανάγκη που υπάρχει για νομικά δεσμευτικό διοντολογικό κώδικα για ε, την άσκηση ε, lobbying στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για το πώς κινούνται οι διάφορες ομάδες πιέσεων, πιέσεων συμφερόντων. Będę Państwa informować o θα σας ενημερώνω ε, για τις εξελίξεις όταν θα έχω νεότερα. Και τώρα ο πρόεδρος Σούλτς έχει ζητήσει το λόγο, όχι. Δεν ζητήσατε το λόγο. Διαδικαστικό, η κυρία Αλφάνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να μιλήσω πριν από εσά για να αναφερθώ στην αποφασιστικότητα αυτού του Κοινοβουλίου να ζητήσει τις την παρέτηση και του άλλου συναδέλφου που δεν έχει υποβάλει την παρέτησή του σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο για όλα όσα αποφάσισε με αποφασιστικότητα και στεναρότητα που θέλει να εφαρμόσει πολιτική μηδενικής ανοχής διότι εκεί υπονομεύεται η αξιοπιστία όλων μας στο Κοινοβούλιο και κυρίως θα πρέπει να θυμόμαστε ότι εκπροσωπούμε 500 εκατομμύρια πολίτες και όχι τα λόμπι. Ε, Σας ευχαριστώ κυρία Αλφάνο. Θα συναντηθώ με τον τρίτο συνάδελφο που δεν έχει παραιτηθεί ακόμα για να συζητήσουμε ακριβώς αυτό το θέμα που θίξατε. Ο συνάδελφος Γκόλνιτς. Κύριε Γκόλνιτς. Κύριε Πρόεδρε, εγκρίνω πολύ την αυστηρότητά σα και ελπίζω ότι θα εφαρμοστεί επίση στους δημοσιογράφους εκείνου που έχουν μια προκλητική συμπεριφορά και πραγματικά κάνουν σοβαρά, σοβαρά σφάλματα. Κατά τα άλλα ισχύεται τεκμήριο αθότητε. Θα ήθελα να σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μάρτιν ζήτησε το λόγο. Συνάδελφε Μάρτιν. Θα ήθελα επίσης ε, θα ήθελα να πω ότι υπερασπίζομαι τους δημοσιογράφους. Θεωρώ ότι είναι αξιόλογο αυτό κύριε Μπούζεκ και ε, πραγματικά θα ήθελα να, οι συνάδελφοι αυτοί να παρετηθούν πριν αποκαλυφθούν οι πράξεις τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ούτως ώστε πραγματικά να αποτραπεί περαιτέρω ζημία για το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Θα ήθελα να το λάβετε υπόψη σας κύριε Πρόεδρε και να το διαβιβάσετε προς όλες τις πολιτικές ομάδες. Κυρία Σένεσεν. Δεν έχετε ανάψει το μικρόφωνο σας. Ε, σα Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην προσφώνησή σα είπατε ότι ομιλούσατε εξ ονόματο του Προεδρείου και εξ ονόματο της πλειοψηφία των μελών του Ευρωκοινοβουλίου. Αυτή είναι η άποψη του συνόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πρόεδρε. Είμαστε κατά των, θεμα... των πραγμάτων αυτών που έκαναν οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Σα ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Σα ευχαριστώ, λέει ο κύριο Πρόεδρε, δεν θα είχα ζητήσει τον λόγο αν δεν είχαμε την πρώτη τελευταία αυτή παρέμβαση που ακούστηκε στην Ολομέλεια. Πιστεύω η μηδενική ανοχή ισχύει για όλα τα μέλη αυτού του σώματος για όλους τους ευρωβουλευτές. Θέλω να θέσω το εξής ερώτημα και παρακαλώ να δοθεί ξεκάθαρη απάντηση. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε πρόεδρε ή ο Γενικός Γραμματέας αυτού του Κοινοβουλίου να το επιβεβαιώσει ότι ο κύριος Ευρωβουλευτής Μάρτιν λόγω ελληματικών καταχωρήσεων, λογιστικών καταχωρήσεων, 160.000 ευρώ πρέπει να επιστρέψει στο Ταμείο του Ευρωκοινοβουλίου, σύμφωνα με άποψη του Ευρωπαϊκού, με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.